Συγγνώμη, μια άλλη πληροφορία θα ήθελα να σας δώσω πρώτα. Οι βελγικές αρχές ε, με ενημέρωσαν για την ανάκληση του κυρίου Ζαν Κλοντ Μπάλκο σε μια θέση που είναι συμβίβαστη με τη θέση του Ευρωβουλευτή με βάση το άρθρο 7 ε, της ε, πράξης για τις καθολικές και άμεσες ευρωεκλογές. Με βάση το άρθρο 4, σημείο 1 του κανονισμού θα ήθελα να σας ενημερώσω για τη διακοπή της θητείας του από τις 16 Ιουλίου του 2009. Επίσης, οι βουλγαρικές αρχές με ενημέρωσαν για την ανέκριση της κυρίας Ρουμιάνα Ζελέβα, η οποία ανέλαβε ε, από στις 27 Ιουλίου καθήκοντα ως ε, Υπουργό Εξωτερικών και θα ήθελα να την συγχαρώ για την ανάλυση των νέων ε, καθηκόντων της. Φυσικά η θέση αυτή είναι ασυμβίβαστη με τη θέση του Ευρωβουλευτού. Με βάση το άρθρο 7 τρίτο εδάφιο της πράξης που αφορά τις ε, άμεσες και καθολικές ευρωεκλογές και το εκτελεστικό άρθρο 4 του κανονισμού από τις 27 Ιουλίου λοιπόν δεν ισχύει πια η κοινοβουλευτική θητεία της ε, κυρίας από τη Βουλγαρία που ανέλαβε ως υπουργό Εξωτερικών. Έχω και διάφορες πληροφορίες. Οι βελγικές αρχές με ενημέρωσαν για την ε, ανάδειξη του κυρίου Μάρκα Ταραμπέλη στην θέση του Ευρωβουλευτού που ε, αντικαθιστά τον κύριο Ζαν Κλοντ Μαρκό με ισχύ από τις 16 Ιουλίου του 2009. Οι βουλγαρικές αρχέ με ενημέρωσαν για την ε, εκλογή ε, ως Ευρωβουλευτή του κυρίου Άντζεϊ Κοβάτσεφ, αντικαθιστώντας την κυρία Ζελέβα, με ισχύ από τις 27 Ιουλίου του 2009. Με βάση το άρθρο 3, δεύτερο εδάφιο του κανονισμού, θα πρέπει να γίνει η ε, εξακρίβωση της εντολής. Εφόσον ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία, οι δύο νέοι ευρωβουλευτές θα αναλάβουν τα καθήκοντά τους ως πλήρη μέλη υπό τον όρο φυσικά της υπογραφής ε, της δήλωσης με την οποία θα δηλώνουν ότι δεν ασκούν κανένα άλλο ε, λειτουργήμα ή επάγγελμα που είναι συμβίβαστο με την ιδιότητα του Ευρωβουλευτού. Ο πρόεδρος ε, των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών με ενημέρωσε ότι ο κύριος Έντουαρτ Μακμίλαν Σκοτ δεν είναι πια μέλος της ομάδας τους από τις 20 Ιουλίου του 2009. Έλαβα από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και των ε, ε, Ευρωπαίων Δημοκρατών καθώς και των Πρασίνων της Ευρώπης για την ε, Ευρώπη των πολιτών ε, μερικά ψηφίσματα σε σχέση με αλλαγές σε κοινοβουλευτικές επιτροπές και ε, διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπίες,